κυρία Πρόεδρος. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Έλαβα εκ μέρου των ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών αιτήσει τροποποίηση στι κοινοβουλευτικέ επιτροπές και στι διακοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείες ο κατάλογος των διορισμών θα δημοσιευθεί στα συνοπτικά πρακτικά αυτής της Συνόδου. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις ως προς την, ένταξη, ε, ως προς την έγκριση των συνοπτικών πρακτικών, οι διορισμοί θα εγκριθούν. Συνεχίζουμε την ημερήσια μας διάταξη, η οποία προβλέπει απόψε την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κύρωση και την εφαρμογή των αναθεωρημένων συμβάσεων τους διεθνούς οργάνους εργασίας. Ε, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες. Το λόγο λοιπόν έχει για τρία λεπτά ο προ... ένας από τους συντάκτες, ο κύριος Σέρκας. Mr. Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζουμε ότι η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική κρίση και οι μελλοντικές προκλήσεις σημαίνουν